του Συμβουλίου και της Επιτροπής όσον αφορά την παρακολούθηση δικηγόρων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Καλίνα Λουκασέφικα, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Uh, uh, uh, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, το Συμβούλιο εκλήθη να παρέμβει σχετικά με το θέμα παρακολούθησης δικηγόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβανόμεθα ότι υπάρχει και προφορική ερώτηση επί του θέματος. Ε, υπευλήθη από τη βουλευτή κυρία Σαρτζεντίνη η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση Ολλανδικής Δικαιογορικής Εταιρείας από τις ε, υπηρεσίες πληροφοριών ενός κράτους μέλους. Καταρχήν να τονίσω ότι η Προεδρία του Συμβουλίου δεν είναι σε θέση να κάνει οδήποτε σχόλιο σχετικά με ισχυρισμούς ότι οι μυστικές υπηρεσίες κρατών μελών μυστικά παρακολουθούν του συνομιλία δικηγόρων και των πελατών τους. Στα πλαίσια της συνθήκη τη Λισαβόνας, η διατήρηση του δικαίου και της τάξεως και η διασφάλιση της εσωτερικής ασφάλειας είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το Συμβούλιο λοιπόν δεν έχει ενημερωθεί για οποιασδήποτε δραστηριότητες παρακολούθησης από εθνικές υπηρεσίες υπεύθυνε για τη διασφάλιση της εθνικής ασφάλειας. Θέλω επίσης να τονίσω ότι η συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τέτοιες υπηρεσίες ασφαλείας εθνικές δεν διέπονται από το ενωσιακό δίκαιο. Ε, η οδηγία του 95 και η απόφαση πλαίσιο του 2008 για την προστασία δεδομένων δεν ισχύουν εδώ η πρόταση της Κομισιόν του 12 για μια οδηγία σχετικά με την προστασία δεδομένων από αρμόδιες αρχές για την πρόληψη, διερεύνηση, αποκάλυψη και δίωξη εγκληματικών δραστηριοτήτων λέει ρητά ότι δεν θα ισχύει δεν θα εφαρμόζεται εις ό,τι αφορά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια μιας δραστηριότητας η οποία αφορά την εθνική ασφάλεια. Για τον ίδιο λόγο η Προεδρία δεν είναι σε θέση να εκφραστεί, να εκφέρει γνώμη σε σχέση με το αν συνάδουν με το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων οι ε, δραστηριότητες αυτές. Η οδηγία σε σχέση με το δικαίωμα πρόσβασης ε, σε δικηγόρο ε, προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη θα σέβονται την εμπιστευτικότητα της επικοινωνίας μεταξύ υπόπτων ή κατηγορουμένων και των δικηγόρων τους κατά την άσκηση του δικαίωματος πρόσβαση σε υπηρεσίες δικηγόρου. Όμως η διάταξη αυτή όπως και όλη η οδηγία ε, είναι το αποτέλεσμα του έργου των εθνικών υπηρεσιών που διασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια σύμφωνα με τις συνθήκες. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρία Γιούροβα, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αξιότιμα μέλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί σε σχέση με το θέμα που προβάλλεται και από τα ΜΜΕ ε, σε σχέση με την παρακολούθηση των δικηγόρων. Το δικαίωμα της ιδιωτικής σφαίρας στην επικοινωνία ε, δικηγόρου ε, πελάτη προστατεύεται από το άρθρο 9 και το δικαίωμα ε, και το άρθρο 47 και 48 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, κεφάλαιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως πρέπει να πούμε ότι ο χάρτης εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν ενωσιακό δίκαιο. Ε, το θέμα της εθνικής ασφάλειας παραμένει η αρμοδιότητα των κρατών μελών. Έτσι λοιπόν, όταν τα κράτη-μέλη αρχίζουν δραστηριότητες μυστικής παρακολούθησης για λόγους εθνικής ασφάλειας, ε, δεν εμπίπτουν στο ενωσιακό δίκαιο. Έτσι λοιπόν ο χάρτης γενικά δεν είναι εφαρμοστέος. Τούτου λεχθέντος η ρήτρα εξαίρεσης θα πρέπει να ε, ερμηνευθεί αυστηρά ε, εις ό,τι αφορά την νομολογία των δικαστηρίων. Οποιοδήποτε κράτος μέλος ε, θέλει να αξιοποιήσει τέτοιες εξαιρεσει, πρέπει να αποδείξει ότι είναι απαραίτητη η προσφυγή σε τέτοια μέσα για να προασπιστούν τα σημαντικά ε, ε, συμφέροντα ασφαλείας. Τα εθνικά συστήματα ε, προβλέπουν ε, τις ανάλογες ε, ρήτρες προστασίας σε αυτή την περίπτωση. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίζεται το δικαίωμα δίκαιη για δίκαιη δίκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό φροντίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από το 2009 έχουμε επιτελέσει σημαντική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση με τη θέσπιση τριών οδηγιών για το δικαίωμα διερμηνίας και μετάφρασης το 2010 για το δικαίωμα στην ενημέρωση από το 2012 και πρόσφατα το δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες δικηγόρου. Η οδηγία για το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο πρέπει να περάσει μέχρι τις 27 Νοεμβρίου του 2016 στην Εθνική Νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει εκ του σε αυτή τη διαδικασία. Το άρθρο 4 της οδηγίας σαφώς αναφέρει την αρχή σεβασμού της εμπιστευτικότητας στην επικοινωνία μεταξύ υπόπτων ή κατηγορουμένων και των δικηγόρων τους όταν εξασκούν, ασκούν το δικαίωμα πρόσβαση σε υπηρεσίες δικηγόρου. Όμως θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι η οδηγία επικεντρώνεται στο δικαίωμα των υπόπτων και κατηγορουμένων προσώπων στις ποινικέ διαδικασίες. Γι' αυτό διευκρινίζεται στις αιτιολογικές σκέψεις ότι η εμπιστευτικότητα αφορά μόνο την πραγματική επικοινωνία κατά την άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης ε, από τον δικηγόρο ενός υπόπτου ή κατηγορουμένου. Δεν αφορά δικηγόρους που ενέχονται σε εγκληματικές δραστηριότητες του ε, υπόπτου ή κατηγορουμένου. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ας περάσουμε στον κύριο Λενάς. Ξεκινάει ο κύκλος των πολιτικών ομάδων. Για 1,5 λεπτό λοιπόν. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Οι σχέσεις δικηγόρου πελατών είναι ιδιαίτερα και το ζήτημα της εμπιστευτικότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες εμπιστεύονται το κράτος δικαίου. Αυτό αποτελεί βασική αρχή της δημοκρατίας. Αυτό από την άλλη όμως δεν σημαίνει ότι κανείς ποτέ δεν μπορεί να συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες ή ότι θα ήταν αδύνατο να συμβεί κάτι τέτοιο. Πιστεύω ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσαμε να δεχθούμε μια τέτοια πρακτική, να διοδοτήσουμε δηλαδή τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά τις σχέσεις ε, δικηγόρων πελατών, αρκεί όμως να ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες και εφόσον δικαιολογούνται από την υπεράσπιση της ασφάλειας μιας χώρας. Η συγκέντρωση τέτοιων ευαίσθητων πληροφοριών μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντική για τα κράτη-μέλη προκειμένου να καταφέρουν να εγγυηθούν την ασφάλεια των πολιτών τους. Πρέπει λοιπόν να δούμε και τη διάσταση αυτή στα πλαίσια αυτή τη συζήτηση που διεξάγουμε. Όπω είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερόμαστε ένα ζήτημα εθνική αρμοδιότητο και η παρακολούθηση δικηγόρων, εφόσον τελικά συνέβη στην Ολλανδία, αποτελεί τελικά ένα εθνικό ζήτημα. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει οι εθνικές αρχές Ολλανδίας ή το Εθνικό Κοινοβούλιο της χώρας να ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Λοπές Αγγιλάρ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστώ την Επίτροπο. Έχω την εντύπωση ότι αυτή η συζήτηση έχει πολύ περιορισμένο θέμα και μάλιστα ίσονος σημασίας ε, σε σχέση με αυτά που απασχολούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό θα έλεγε κανείς αν μας άκουγε. Όμως θα είχε λάθος, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα. Μιλούμε για υπονόμευση δικαιωμάτων, ελευθεριών, για πλήγμα στην ιδιωτικότητα των συνομιλιών, αλλά και για πολύ μεγάλο πλήγμα ε, στις, ε, στους συνηγόρους και στην εκπροσώπηση και υπεράσπιση ενώπιον της δικαιοσύνης του οποιοδήποτε. Μιλούμε για ε, οικουμενική καθολική κατασκοπία ουσιαστικά από ε, τον εξοπλισμό και τα μέσα των κρατών μελών, τα οποία είναι εξαιρετικά προηγμένα και εξελιγμένα. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να το αρνηθούμε αυτό, να πούμε όχι, να πούμε ότι θα τα παρεμποδίσουμε με τη Χάρτα Θεμελιωτών Δικαιωμάτων, με τη Συνθήκη της Λισαβόνας, με τη ε, νομιμοποίηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο είναι συνομοθέτης. Όλα αυτά θα κραδένουμε όταν θα διώκουμε και θα τιμωρούμε το, την διασυνοριακή σοβαρή εγκληματικότητα ε, η οποία πλήττει το δικαίωμα στην υπεράσπιση, το δικαίωμα να έχει κανείς δικηγόρο, ε, το δικαίωμα να ε, τη χάνει προστασίας σε περίπτωση δικαστικών διώξεων. Ε, από πλευράς λοιπόν κοινοβουλευτικού ελέγχου έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την υποχρέωση να απαιτήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να νομοθετήσει, να προτείνει νομοθετία για ε, αυτό το θέμα έτσι ώστε να ε, πάνε τα πράγματα καλύτερα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βίξτρομ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι σημαντικό στο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, στα ευρωπαϊκά κράτη όπου επικρατεί το κράτος δικαίου είναι το δικαίωμα να μιλά κανείς ελεύθερα με το δικηγόρο του, να έχει ένα νόμιμο εκπρόσωπο και όλοι οι, όλες οι συνταγματικές προβλέψεις για την κατοχήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων το ε, περιλαμβάνουν αυτό σαφέστατα. Τώρα, οι πληροφορίες που ανταλλάσσονται μεταξύ πελάτη και δικηγόρου, εάν διαραίουν, αυτό σημαίνει ότι έχει υπονομευθεί, έχει καταστρατηγηθεί αυτό το δικαίωμα και αυτό είναι απαράδεκτο. Από ό,τι φαίνεται, παρακολουθούσε το δικαστή Ντάκτη Ριβιέρα η Ολλανδική Υπηρεσία Πληροφοριών και έχουμε και σχετικά παραδείγματα σε άλλα κράτη-μέλη. Θέλω απάντηση στο ερώτημά μου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θεωρούν ότι αυτού του είδους η κατασκοπία σε δικηγορικές εταιρείε αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, ναι ή όχι, ευθυγραμμίζεται με τη συνθήκη, με τη χάρτα, με όλα τα δικαιώματα τα οποία απολαμβάνουμε βάσει αυτών των κειμένων εμείς οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ποια είναι επιτέλους η άποψη ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου. Αυτό έγινε γιατί μπαίνει στο πλαίσιο της ε, εθνικής ασφάλειας. Ε, τότε πώς ορίζεται την εθνική ασφάλεια. Αυτό σημαίνει ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας κάθε φορά μπορεί να στερούνται πολίτες των δικαιωμάτων τους και να μην έχουν κανένα τελικά ποια μέτρα θα θεσπίσει το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα, το απόρριτο στις συνομιλίες μεταξύ δικηγόρων των και πελατών. Θα λάβετε συγκεκριμένα μέτρα εναντίον των χωρών μελών. Πότε θα επανέλθετε με αποδεκτό επιτέλους ορισμό της έννοιας εθνική ασφάλεια ο κύριος Χουαρίστη Αμπαούντς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας μιλήσω για τη κατάσταση στη χώρα μου, τη χώρα των Βάσκων. 16 πολίτες συνελήφθησαν χθε από την ε, χώρο φυλακή. Δικηγόροι που υπερασπίζονται Βάσκους κρατουμένους. Και μεταξύ άλλων και άλλωστε 35 ε, βάσκοι κατηγορούμενοι θα ε, δικάζονταν χθες στη Μαδρίτη. 85.000 ε, άνθρωποι διαδήλωσαν στο Μπιλμπάο για τις συνθήκες κράτησης στις φυλακές. Τελικά η αστυνομία έψαξε ε, τους χώρους ενός συνδικάτου και πήρε τα χρήματα που είχε συγκεντρώσει το συνδικάτο από τους συμμετέχοντες στην πορεία. Ουσιαστικά συνελήφθησαν αυτοί οι άνθρωποι γιατί εργάζονται στον χώρο της δικαιοσύνης. Είναι απαράδεκτο ένα κράτος μέλος να καταστρατηγεί τέτοιου είδους θεμελιώδη δικαιώματα και μάλιστα με τέτοια τιμωρησία. Είναι απαράδεκτο ένα κράτος μέλος να απορρίπτει ε, την ευρωπαϊκή νομοθεσία υποτίθεται για να ε, υπάρξει εσωτερική ασφάλεια ενώ ήδη εκτίονται οι ποινές. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, αυτό είναι εκδίκηση και θα πρέπει να γίνει συζήτηση με τη διαδικασία του καταπήγοντος. Είναι θέμα δικαιωμάτων. Το Ισπανικό κράτος δείχνει ότι δεν είναι καθόλου δημοκρατικό και το μόνο που κάνει είναι να, να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από το κράτος, ε, ε, από το κράτος δικαίου. Καλό την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ισπανικό κράτος να κάνουν σωστά βήματα για να επιληθεί η σύγκρουση. Η βασική κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Ευχαριστώ. Δεν έχετε άλλο χρόνο κύριε, λέει η κυρία Πρόεδρος. Η κυρία Σαρτζεντίνη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές να είναι πιο διαλλακτικές, να δείχνουν εμπιστοσύνη, να επιβάλλουν τον νόμο. Αλλά βλέπουμε τελικά ότι στην πράξη δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο πολλές φορές. Ήταν θέμα χρόνου τελικά, προτού προκύψει ένα τέτοιο ζήτημα σε αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα όπου αναφερόμαστε βασικά σε παρακολούθηση και δικηγόρων στην Ολλανδία. Οι Ολλανδικές Μυστικές Υπηρεσίες AIVD παραδέχθηκαν ότι όντως παρακολουθούσαν τις τηλεφωνικές συνομιλίες του δικηγορικού γραφείου Πράκεν Ντολιβέιρα. Αν αποδεχθούμε κάτι τέτοιο για τους δικηγόρους, τι θα γίνει με άλλα επαγγέλματα όπου χρειαζόμαστε υψηλό βαθμό εμπιστευτικότητας, όπως για παράδειγμα το ιατρικό επάγγελμα. Η οδηγία του 2013 όσον αφορά τα δικαιώματα των δικηγόρων στο άρθρο 4 λέει ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπερασπιζόμαστε την εμπιστευτικότητα της σχέσης δικηγόρου-πελάτη. Σε κάποιο άλλο άρθρο επίσης οδηγίες αυτής αναφερόμαστε στο δικαίωμα της δίκαιης δίκης. Απευθύνομαι λοιπόν και στον κύριο Τίμερμαντς, που δεν είναι εδώ βέβαια αλλά και σε εσά κυρία Γιούροβα προκειμένου να δώσετε μία απάντηση στο προφορικό μας ερώτημα. Τι θα κάνετε προκειμένου να επιβληθεί το κοινοτικό δίκαιο και προκειμένου οι Ολλανδικές αρχές αλλά και οι υπόλοιπε εθνικές αρχές να σέβονται τελικά τον εμπιστευτικό χαρακτήρα της σχέσης δικηγόρου-πελάτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Επαναλαμβάνομαι βέβαια, αλλά είναι αλήθεια. Η σχέση δικηγόρου-πελάτη στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Και η προστασία αυτή της εμπιστευτικής σχέσης ε, πρέπει να καλύπτει όχι μόνο δικηγόρους αλλά και δημοσιογράφους και γιατρούς και άλλους επαγγελματίες. Είναι ένα βασικό στοιχείο αυτό κάθε δημοκρατίας και κάθε κράτος μέλους λοιπόν ως πολιτικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση εμείς καλούμεθα να θεωρήσουμε αυτό το στοιχείο ως πυλώνα της ένομης τάξης. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται εδώ για μεμονωμένη περίπτωση που στον τομέα ασφαλείας παίζει σημαντικό ρόλο και σε αυτή την ιδιαίτερη περίπτωση σκέπτομαι ότι ε, ε, ίσως ε, εδώ υπάρχουν κάποιες περιορισμένες αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λάβουμε και αυτό υπόψη, γιατί πρόκειται για θέματα ασφαλείας. Είναι περιορισμένες οι αρμοδιότητες και η εθνική ασφάλεια είναι πρωτίστως αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το Συμβούλιο δεν μπορεί να δράσει σε επίπεδο κράτους μέλους ή να, να, να, κινήσει διαδικασία. Εδώ υπεύθυνη είναι η δικαιοσύνη, το Υπουργείο Εσωτερικών στην Ολλανδία και νομίζω ότι η Ολλανδία είναι αρκετά δημοκρατικό κράτος ούτως ώστε να το διερευνήσει το θέμα. Και δεν είναι κράτος που παρακολουθεί τους πολίτες. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος Άλμπρακτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι θα πρέπει να συζητήσουμε δύο ζητήματα. Πρώτον, δεν είναι η μόνη και πρώτη περίπτωση όπου ένα κράτος μέλος κρύβεται πίσω από τις λεγόμενες εξαιρέσεις όσον αφορά την εθνική ασφάλεια στα πλαίσια των συνθήκων, ξέρουμε ότι και η Βρετανική Υπηρεσία Μυστικών Πληροφοριών κατέστρεψε πληροφορίες που είχαν σχέση με δημοσιογράφους, παρακολουθήσεις δηλαδή δημοσιογράφους, αυτή τη στιγμή ακούμε όλο και περισσότερο για παρακολουθήσεις δικηγόρων, όπου προβάλλεται το πρόσχημα της εθνικής ασφάλειας. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά να ζητήσει από τα δικαστήρια να της δώσουν ένα συγκεκριμένο ορισμό για το τι σημαίνει εθνική ασφάλεια και σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιείται αυτό το επιχείρημα, αυτό το πρόσχημα. Δεύτερον, η παρακολούθηση δικηγόρων και η παρακολούθηση δημοσιογράφων τι ακριβώς σημαίνει, σε τι συνίσταται. Όσον αφορά τους δικηγόρους, τουλάχιστον μετά τις επιθέσεις της προηγούμενης εβδομάδας βλέπουμε ότι ενδεχομένως να επεκταθούν δραστηριότητες παρακολούθησης τόσο στους δικηγόρους όσο και στους δημοσιογράφους. Πρέπει λοιπόν να δούμε με ποιο τρόπο θα συλλέγονται αυτά τα δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρία άτομα για το Catch the Eye, ο κύριος Πόλτσακ πρώτος, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, Κυρία Υπουργέ, δεν μπόρεσα να μιλήσω για το ζήτημα των ποσοστώσεων, αλλά θα το, μάλλον κάποιων αναφορών που γίνανε. Η κυρία Υπουργός αναφέρθηκε στον χάρτη, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, όπου λέγεται ότι ε, το ζήτημα αυτό το οποίο συζητάμε σήμερα μπορεί να καλυφθεί από το ενωσιακό δίκαιο. Τι γίνεται όμως με τα κράτη-μέλη εκείνα τα οποία δεν έχουν μεταφέρει ακόμα στην εθνική τους νομοθεσία το εν λόγω δίκαιο. Συγκεκριμένα, αν ένα κράτος μέλος παραβιάσει την εν λόγω νομοθεσία, ποιος μπορεί να το υποχρεώσει τελικά να συμμορφωθεί με τον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, ποιος μπορεί τελικά να επιβάλλει κυρώσεις σε αυτό το κράτος μέλος. Πρέπει να μας απασχολήσει αυτό, γιατί η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ δικηγόρου πελάτη είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραβιάζεται. Τι θα γίνει αν δεν νομοθετήσουμε για το ζήτημα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε πάρα πολλούς τομείς τίθεται ένα αμφιβόλο η σχέση δικηγόρου-πελάτη. Αυτό το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, συγκεκριμένα με κάποιους βάσκους κρατούμενους, Επίσης είδαμε ότι έχουν γίνει παρακολουθήσεις ακόμα και σε γραφεία συνδικαλιστικών οργανώσεων. Νομίζω ότι όλοι συμπεριλαμβανομένων των δικηγόρων θα πρέπει να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμά τους χωρίς εκφοβισμό, χωρίς παρακολουθήσεις. Δυστυχώς στην Ιρλανδία ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι μπορεί να συμβεί όταν το κράτος εμποδίζει τελικά τους δικηγόρους από το να επιτελούν το έργο τους η δολοφονία δικηγόρων στην Ιρλανδία στο παρελθόν με τη βοήθεια και την υποκίνηση των Βρετανικών αρχών καταδεικνύει τελικά ακριβώ την τραγωδία στην οποία μπορούμε να καταλήξουμε αν τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προασπίζει τα σχετικά δικαιώματα δικηγόρων πελατών. Ο κύριος Κοράο, τελευταίος ομιλητής για ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ δεν συμφωνώ με τον κύριο Λένερτς, ο οποίος είπε ότι μέσω του προφορικού αυτού ερωτήματος τελικά καλύπτουμε ένα ζήτημα που δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ θεωρώ, όπως είπε και η κυρία Σαρτζεντίνο, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω ότι τελικά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να εθελοτυφλούμε μπροστά σε κάποια βασικά δικαιώματα όπως το δικαίωμα υπεράσπισης, το δικαίωμα δίκαιης δίκης, το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα, τα οποία προκειμένου να προασπίσουμε ή να νομοθετήσουμε για αυτά, απαιτήθηκε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να τηρήσουμε τι διατάξει τι οποίε έχουμε ήδη εγκρίνει. Έχουμε μία οδηγία του 2003, η οποία πρόδειλα παραβιάζεται αυτή τη στιγμή. Τα όσα συμβαίνουν στο Ολλανδία θα μπορούσαν αύριο μεθαύριο να συμβούν σε οποιαδήποτε χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει λοιπόν συγκεκριμένα να τοποθετηθεί τόσο το Συμβούλιο όσο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κυρία Γιούροβα έχει το λόγο εξ ονόματο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρίε και κύριοι, συμφωνώ ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό, αλλά και πάλι πρέπει να επαναλάβω ότι αυτή τη στιγμή το θέμα είναι στη δικαιοδοσία των κρατών μελών. Εμείς έχουμε θεσπίσει κανόνες για την παρακολούθηση, αλλά εδώ πρόκειται για εθνικές υπηρεσίες ασφαλείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να παρακολουθήσει την εφαρμογή της οδηγίας για το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο, που, όπως είπα, ενσαρκώνει την αρχή του σεβασμού της εμπιστευτικότητας ε, ε, στη σχέση μεταξύ υπόπτων κατηγορουμένων και των δικηγόρων τους. Ε, αυτοί έτσι έχουν τώρα τα πράγματα. Οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρακολουθήσει από κοντά τις εξελίξεις στο θέμα αυτό και σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο συμπεριλαμβανομένων σχετικών υποθέσεων ε, που τη χειρίζεται το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Καλνίνα Λουκασέβιτσα, εξ ονόματος του Συμβούλιο. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ε, ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές για τα θέματα που έθεσαν, για τις ανησυχίες που εξέφρασαν κατά τη διάρκεια αυτή, αυτής της συζήτησης. Θα διασφαλίσω ότι το Συμβούλιο θα ενημερωθεί για τη συζήτησή μου μαζί σας. Θα τα μεταφέρω όλα αυτά. Το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει αυτό το συγκεκριμένο θέμα που μας απασχολεί και δεν έχει οθετήσει θέση επ' αυτού για λόγους που σας έχω ήδη εξηγήσει. τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, θέσουν τους δικούς τους ε, κανόνες ε, για θέματα εθνικής ασφάλειας. Σας ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σας αλλά και για την καλή συζήτηση που είχαμε. Η Πρόεδρος.